που είναι η έκθεση της κυρίας Σίλβια Ιβόν Κάουφμαν σχετικά με τον ενιαίο τύπο θεωρήσεων. Θα παρακαλέσω πρώτα λοιπόν την εισηγήτρια να μιλήσει και έχει στη διάθεσή της τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εσείς κυρία Επίτροπε. Ήδη από το 1995 υπάρχει ενιαία διαμόρφωση του ε, διαμόρφωση της θεώρησης ενιοτύπου. Εξακολουθούν όμως να απαιτούνται έγγραφα σε μορφή χαρτιού. Δεν ε, σημειώνονται όλα τα δεδομένα ηλεκτρονικά και χωρίς δυνατότητα χρήση ηλεκτρονικών μέσων πρέπει οι συνοριοφύλακες να μπορούν να ε, διαπιστώνουν τη γνησιότητα του εγγράφου που τους τίθεται υπόψη. Το η φυστάμενη αντίληψη περί ασφάλειας είναι παραπάνω από 20 χρόνια ε, παλαιά και έχει βελτιωθεί, έχει ε, τροποποιηθεί δύο μόνο φορές έως τώρα. Οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές ανάγκες ασφαλείας. Δηλαδή, οι θεωρήσεις που εκδίδονται τώρα δεν είναι ασφαλείς απέναντι σε παραχαράξεις και πλαστογραφήσεις και έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά πολλά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα κενό ασφαλείας που πρέπει να αρθεί. Με τη σημερινή μας ψηφοφορία θα δώσουμε πράσινο φως για ένα νέο σχεδιασμό των θεωρήσεων που θα είναι δεσμευτικό για τις χώρες μέλη. Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει επεξεργαστεί τις ε, νέες ε, διατάξεις ασφαλείας με νέους τρόπους εκτύπωσης και με λεπτομέρειες που θα δυσκολέψουν πάρα πολύ το έργο των παραχαρακτών στο μέλλον. Παράδειγμα, ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας μπορούσαν έως τώρα να αποκόπτονται. Τώρα αυτό όμως δεν θα είναι δυνατό στο μέλλον, διότι θα βρίσκονται ακριβώς στο μέσον του σήματος. Η Κομισιόν τον Ιούνιο του 2015 είχε υποβάλει πρόταση. Η έκθεσή μου ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία ε, πέρσι από την Επιτροπή θεμελιώδων Ελευθεριών το 2016 δηλαδή. Και τον Απρίλιο φέτος μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε επιτέλους τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών. Και εκφράζω την ικανοποίησή μου ιδιαίτερω διότι έχουμε επιτέλους μια νομικά ασφαλή λύση για να μπορέσει να συμμετάσχει και η Ιρλανδία παρόλο που δεν αποτελεί μέρος του χώρου Σέγγεν. Δεν θα ήθελα να αποκρύψω ωστόσο ότι θα προτιμούσα να είναι συντομότερη η μεταβατική περίοδος όπου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι μέχρι τώρα ισχύουσες προξενικές θεωρήσεις. Βεβαίως, οι προκηρύξεις για την τύπωση των νέων θεωρήσεων και η παραγωγή και η διανομή τους σε όλα τα προξενία πανταχού του κόσμου χρειάζονται χρόνο. Οι 15 μήνες ως ανώτατο όριο είναι ωστόσο αρκετά μακρά περίοδος και είναι βέβαια και το απότατο όριο που μπορούσαμε να αποδεχθούμε. Ελπίζουμε ότι οι χώρες μέλη δεν θα εξαντλήσουν την μεταβατική αυτή περίοδο και θα κλείσουν το δυνατόν συντομότερο το κενό ασφαλείας υιοθετώντα και εισάγοντα τι νέε προξενικέ θεωρήσει. Ολοκληρώνοντα, κυρία Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω τι σκιώδει συγγήτριε και συγγητέ των άλλων πολιτικών ομάδων για την πολύ θετική συνεργασία καθώς επίσης ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως την Μαλτέζικη Προεδρία, διότι η συμφωνία που επετεύχθη δείχνει ότι θέλουμε όλοι, έχουμε όλοι κοινό στόχο την αύξηση της ασφαλείας στην Ευρώπη και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αξίζει κάθε προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κάουφμαν. Θα προσκαλέσω τώρα την Επίτροπο κυρία Μάρμστρομ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πρώτα την εισηγήτριά σα, κυρία Κάουφμαν, για το έργο που επετέλεσε, καθώ και τι κοιόδη εισηγήτριε και εισηγητέ. Βεβαίω ήταν μακρά η διαδικασία, αλλά όμω σημαντική. Η εγγύηση τη ασφαλεία των εγγράφων ταξιδιού είναι πολύ σημαντικό παράγον για την καταπολέμηση των παραχράξεων προστασία των συνόρων, εξασφάλιση τη εσωτερική ασφάλεια και καλύτερη διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Χαίρομαι λοιπόν για το νέο τύπο κοινών, ε, για τον νέο κοινό μάλλον τύπο, νέο τύπο θεωρήσεων. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση το 2015, έγινε αυτό για να υπάρχουν νέες ετικέτες επισήμανσης επί των προξενικών θεωρήσεων που θα είναι ασφαλής απέναντι σε προσπάθειες παραχάραξης. Πρόκειται για μέρος μιας συνολικότερης προσέγγισης για την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριων, ε, αδειών παραμονής και βεβαίως και με την χρήση βιομετρικών δεδομένων. Πράγματι πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια μέχρι ότου καταλήξουμε σε συμφωνία και ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σκληρή δουλειά υπό την ηγεσία βεβαίω και κατεύθυνση της κυρίας Κάουφμαν. Ε, Χρειάζεται πλέον οπωσδήποτε να προχωρήσουμε Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει πολύ σύντομα, ώστε η εισαγωγή του ενιαίου τύπου προξενικής θεώρησης να συμβάλλει στην αύξηση της εσωτερικής ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και πέρα τώρα στον κύριο Τζαμπάσκη από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, συνάδελφοι. Ο συντάκτης γνωμοδότησης ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ε, με απειλή της ασφάλειάς μας από την τρομοκρατία είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν ε, σημαντικά και συνεπή μέτρα. Και το μοντέλο ενιαίας θεώρησης, θεώρηση ενιαίου τύπου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αύξηση το, της πλαστογράφησης αυτών των αυτοκόλλητων ετικετών στις θεωρήσεις και είναι όλο και πιο εφάνταστοι οι εγκληματίες που παραχαράσουν ή παραποιούν τέτοιες θεωρήσεις. Επίσης είχαμε αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων ε, και υπάρχει κίνδυνος ε, και νέων τέτοιων τρομοκρατικών επιθέσεων, ε, ιδιαίτερα όταν επιτρέπεται ή γίνεται δυνατή η κυκλοφορία πλαστογραφημένων θεωρήσεων. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε τα σύνορά μας και το μοντέλο θεώρηση νέου τύπου είναι ένα σωστό βήμα προς την καλή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Κοέλιο τώρα για 2,5 λεπτά. Περνάμε στου ομιλητέ από τι ομάδε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε Μάλμστρομ. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την κυρία Κάουφμαν για την ε, εξαιρετική και πολύ αξιόλογη εργασία της και αυτή τη γνώμη εστερνίζεται και ο κύριος Πέτρη Σάραβαμα, που ήταν ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ. Το 1995, όταν καθιερώσαμε τη θεώρηση νέου τύπου, συμπεριλάβαμε στην κοινοτική σφαίρα μια πολιτική που αρχικά εφαρμοζόταν από τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν στο χώρο Σέγγεν. Η ομοιογενοποίηση αυτής της πολιτικής ήταν και εξακολουθεί να μένει σημαντική για, το χώρο της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η θεώρηση είναι μια έγκριση που επιτρέπει την νόμιμη διέλευση ενός εξωτερικού συνόρου και εξασφαλίζει στον κάτοχό της το δικαίωμα να παραμείνει στην επικράτειά μας. Για το χώρο Σέγγεν, η, τα εξωτερικά σύνορα, παρά, παρόλο που νομικά εξακολουθούν να είναι εθνικά σύνορα, στην πράξη είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Η διασφάλισή τους λοιπόν και η αυθεντικότητά τους συνιστά μια ευρωπαϊκή πολιτική και θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητά μας. Το Σέγγεν απαιτεί ευρωπαϊκές πολιτικές που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία του και εξασφαλίζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Το Σέγγεν σημαίνει διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, σημαίνει κοινή πολιτική του ασύλου, πολιτική των θεωρήσεων, πολιτική των επιστροφών, αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία και σημαίνει και σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι τα πλονεκτήματα του χώρου Σέγγεν το οδήγησαν την Ιρλανδία που δεν είναι ε, μέλος του Σέγγεν να ζητήσει συμμετοχή στον κανονισμό. Και μάλιστα τις εποχές που πολλές χώρες ε, προτιμούν να μένουν απ' έξω, όταν διαπιστώνουν τα θετικά αποτελέσματα και τις συνέπειες ζητούν να συμμετέχουν και αυτές σε μερικούς κανονισμούς. Είναι σημαντικός ο κανονισμός, ιδιαίτερα υπό το φως της αύξησης της παράτυπη μετανάστευσης και του εγκλήματος, γιατί τον τελευταίο καιρό είχαμε αύξηση του αριθμού των πλαστογραφήσεων και των παραποίησεων, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συνόρων μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, Χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό και χάρη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγχαρητήρια και πάλι στην κυρία Κάουφμαν και χάρη στη συνδρομή και τη Μαλτέζικη Προεδρία αλλά και τη Αρμόδια Επιτρόπου, ε, ορίμασε η κατάσταση για να εγκρίνουμε επιτέλου τον κανονισμό. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα γιατί πιστεύω ότι έτσι τα σύνορά μα θα είναι πιο ασφαλή. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κινίτσι για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κάφμαν και τους κοιόδες συγητές όλους γιατί εργάστηκαν ε, σκληρά για αυτό το θέμα το οποίο αφορά την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Αυτός ο ενιαίος τύπος θεώρησης των τελευταίων 20 ετών αποτελεί ένα εργαλείο πάρα πολύ βασικό ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων. Παρ' αυτά βλέπουμε ότι συνέχεια έχουμε περιπτώσεις παραχάραξης και απάτης σε πολλά κρατημέλη. Επομένως για αυτό έπρεπε να παρέμβουμε τόσο ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση για περισσότερη ασφάλεια των συμπολιτών μας και να υπάρχει καινούριο τύπος ε, θεώρησης πιο σίγουρος και τεχνολογικά να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που έχουν ε, αναδεθεί. Και επομένως αυτό ήταν μια αντίδραση ξεκάθαρης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπονηθεί η παραχάραξη. Αυτό ήταν βασικό γιατί έχουμε αύξηση των αιτήσεων θεωρήσεων ε, και έχουν αυξηθεί άλλωστε και οι μεταναστευτικές ροές. Και έτσι τώρα έχουμε αυτό τον ενιαίο τύπο θεώρηση με περισσότερα χαρακτηριστικά ασφάλεια, να είναι αυτό το αυτοκόλλητο πιο ε, ασφαλέ, να μην μπορεί να γίνει παραποίηση και να καταπολεμήσουμε την λαθρομετανάσταση ε, και αυτούς που διαμένουν στην επικρά τι μας πέραν του όσο τους επιτρέπεται και των όσων προβλέπει η θεώρησή τους. Οπότε η παραχάριξη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα από το οργανωμένο έγκλημα. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο τώρα ε, στηρίζονται και τρομοκρατικές οργανώσεις. πρέπει έτσι να ελέγξουμε καλύτερα τα σύνορα και έτσι να ελέγχεται ποια είναι τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Είναι θέμα εσωτερική ασφάλεια επίση και πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα και να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση του συστήματο θεωρήσεων. Σα ευχαριστώ για τη δουλειά σα, συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Τόμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι σύγχρονε τεχνολογίε δυστυχώ διευκολύνουν τη ζωή όχι μόνο των ομοταγών πολιτών, αλλά και εκείνων που εσκεμμένα παρακάμπτουν του νόμου. Το οργανωμένο έγκλημα πολύ συχνά είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πολλέ φορέ φορές προηγείται ένα-δύο βήματα των αρχών ασφαλεία. Η πλαστογράφηση των θεωρήσεων είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και χαιρετίζω την πρόταση κανονισμού που πραγματικά συνιστά βήμα προόδου και προστατεύει του Ευρωπαίου πολίτε ε, και συμβάλλει στην καλύτερη πολιτική συνεργασία. Αλλά η συνεργασία μα δεν πρέπει να αφορά μόνο του αλλοδαπού πολίτε που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του δικού μα υπηκόου που ταξιδεύουν εκτό Ευρώπη Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι όλοι υπήκοοι των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαλλάσσονται από θεώρηση για τι Ηνωμένε Πολιτείες. Και αυτό είναι ένα είδο διακριτική μεταχείριση. Δεν πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε πολίτε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Θα πρέπει να διευθετήσουμε αυτό το, σύντομα, το θέμα το συντομότερο δυνατό. Δύο λεπτά ο κύριος Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζει η πολιτική μας ομάδα τη θέπιση αυτού του καινούργιου τύπου θεώρησης όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών και συγχαρητήρια για τη δουλειά της στην εισηγητρία. Είναι αλήθεια ότι είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, παραποίησης και αφορούσαν αυτά τα αυτοκόλλητα πολλών κρατομελών, αλλά επίση έτσι οι εμπειρογνώμονε είπαν ότι έτσι όπω έχει αυτό το πρότυπο που ισχύει σήμερα δεν ε, αρχή. Και επομένω θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτέ όλε τι απάτε και οπότε έτσι επιφέραμε κάποιε βελτιώσει. Οπότε χωρί ε, επιφύλαξη ε, εγκρίνουμε αυτό που κάνετε κυρία εισηγήτρια. Και έχουμε όμω αυτού του 15 μήνε που είναι μεταβατική περίοδο. Αυτή νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μακρά όμως υπερβολική και επίσης δυστυχώς κάποιου νομικού προβλήματος ε, παρατάθηκε η εκπόνηση αυτής της ε, έκθεσης. Ήταν το πρόβλημα την Ιρλανδία. Οπότε με την ευκαιρία θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή για δύο θέματα κυρία Επίτροπε. Ε, Δημών για όλη την Επιτροπή τα λέω αυτά ότι η κάλυψη των εθνικών θεωρήσεων στο σύστημα πληροφοριών που αφορά τις θεωρήσεις είναι κάτι τόσο σωστό για να καταπολεμηθεί η παραχάραξη σε αυτόν τον τομέα και έτσι θα αναβαθμιστεί η ασφάλεια όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Δεύτερον, δεν θεωρείται ε, ότι θα έπρεπε επίσης να προβλέπεται ένας ενιαίος τύπος για τις ταυτότητες και επομένως ε, όσοι ηθαγενείς ε, τρίτων χωρών κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ένα, μια τέτοια ταυτότητα. Αλλά είναι κάτι που δεν το έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλές φορές ζητούνται 27 διαφορετικές Έχουμε το 27 διαφορετικές ε, ταυτότητες και αυτό βεβαίως φέρνει σύγχυση όσον αφορά τους νοριοφύλακες και ωφελεί ε, τις ε, μαφίε. Οπότε, κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να αναλάβετε σοβαρή πρωτοβουλία ως Επιτροπή για αυτό το θέμα. Η κυρία Βαλέρο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Κάουφμαν και τους υπόλοιπους και οδησηγητές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Πρόκειται για ένα θέμα που διαπιστώνω ότι μας βρίσκει εν γέννη σύμφωνος. Το ισχύον σύστημα ισχύει εδώ και 20 χρόνια και στο μεταξύ έχουν αλλάξει πολλά. Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μεταξύ άλλων κάτι που διευκολύνει και τους παραχαράκτες που πλαστογραφούν τις παλιές θεωρήσεις. Το νέο, ο νέος τύπος, ο νέος τύπος θεώρησης πραγματικά συνιστά ένα βήμα πρόοδου. Το παλιό σύστημα ήταν από το 1995. Ε, θεωρούσαμε τα μόνο τεχνικό, αλλά έχει γίνει πια πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα μετά το, φως, μετά το Brexit. Είναι σημαντικό σήμερα περισσότερο από ποτέ να καταπολεμήσουμε τις πλαστογραφημένες θεωρήσεις και είναι ένα πρόβλημα που διαπιστώνουμε σε πολλές χώρες μέλη. Γι' αυτό και θα πρέπει να εγκρίνουμε μία εναρμόνιση ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της θεωρής ενιαίου τύπου. Σήμερα υπάρχουν κάποιες ε, τεχνολογικές εξελίξεις ε, που λαμβάνουν χώρα ραγδαία, θα πρέπει να τις ε, παρακολουθήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε και γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα θα υπερψηφίσει αυτή την πρόταση προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παλαιστογραφία και την παραχάραξη το συντομότερο δυνατό. Επίσης να μην ε, ε, εμβλακούμε σε μόνο πολιτικά θέματα γιατί υπάρχουν και τεχνικά. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι το αντικείμενο του σημερινού κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων ε, του χώρου Σέγγεν δεν αρκούν πλέον. Και γι' αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η παραχάραξη και η εξού και η νομοθεσία για τον ενιαίο τύπο θεώρησης Σέγγεν. Η χώρα μου δεν συμμετέχει στην, ε, στο χώρο Σέγγεν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεχωριστό σύστημα και ευτυχώ η πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν, τουλάχιστον επίσημα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειάζεται να σφίξουν λίγο τα πράγματα για την παράνομη μετανάστευση. Όποιο βέβαια περάσει τη Μεσόγειο πάνω σε μια βάρκα θα φτάσει και στην Ευρώπη και θα γίνει δεκτός, είτε έχει χαρτιά είτε όχι. Και οι διακινητέ ανθρώπων τους βάζουν μόνο τόση λίγη βενζίνη μέσα στις ε, ε, βάρκες αυτές ώστε να φτάσουν στο ανοιχτό πέλαγος για να μπορέσουν να διασωθούν. Έχει γίνει στην πραγματικότητα όχι πια υπηρεσία διάσωσης αλλά υπηρεσία ταξί για τους παράνομους μετανάστες. Το πόσο σημαντικός είναι ο χώρος Σέγγεν για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό αποδεικνύεται ότι είναι μαγνήτης για τους παράνομους μετανάστες. Αυτή τη στιγμή μπει μέσα στο χώρο Σέγγεν μπορεί να πάει πλέον όπου θέλει και παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί μέρο του χώρου Σέγγεν, θεωρώ ότι η συνοριακή μα έλεγχη είναι πάρα πολύ χαλαρή και ένα πραγματικό χάος. Δείτε τα επίσημα νούμερα μετανάστευσης. Το 2016 273.000 ε, επισήμως όμως 825.000 αριθμοί κοινωνικών ασφαλίσεων χορηγήθηκαν σε άλλο δαπούς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια τεράστια διαφορά. Μια γερμανική ε, μελέτη λέει ότι περιμένουν ακόμα 6 εκατομμύρια μετανάστες να έλθουν στην Ευρώπη. Εμείς οι βουλευτές του UKIP θα απόσχουμε και καλή τύχη για να φτιάξετε το σύστημα θεωρήσεών σας γιατί πάνω θα σας χρειαστεί. 1,5 λεπτό εν Obermeier, κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τύπος θεώρησης είναι σαφές ότι είναι σκόπιμο ώστε να υπάρχουν όλα τα σχετικά δεδομένα και για το ταξίδι προς την Ένωση και για την επιστροφή. Θα πρέπει η χώρα μέλος να γνωρίζει ποιος έρχεται. Αυτό σημαίνει ασφάλεια. Όμως στην, ε, στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να λησμονείται και το ερώτημα ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προξενικής θεώρησης και αυτοί έχουν δυνατότητα να παραμείνουν 90 ημέρες και μετά πρέπει να αποχωρήσουν. Πρέπει και αυτό να συζητηθεί. Φέτος Ουκρανία και Γεωργία εντάχθηκαν και αυτές στον όλο και μακρότερο κατάλογο των χωρών όπου δεν ισχύουν προξενικές θεωρήσεις. Και τώρα έχουν και άλλους υποψηφίους, το Κόσοβο και η Τουρκία. Άρα αυτή η τάση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνεται διαρκώς λησμονεί τις ανάγκες ασφαλείας και φοβούμε ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση στο μέλλον. Θα πρέπει να γίνει συγκεντρωτική η ε, χορήγηση των ε, θεωρήσεων και αυτό θα σημαίνει όλο και περισσότερη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Τζέιμς, ένα λεπτό. Καλημέρα. Πάνω από 20 χρόνια υπάρχει αυτή η πολιτική, όμως δεν είναι πλέον ασφαλής και επιτρέπει πολλές ε, απειλές να αναπτύσσονται σε βάρος των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφάλεια κατά της παραχάραξης και πλαστογράφησης δεν έχει αποτύχει σε πολλές χώρες μέλη και αυτά τα λέει και η ίδια η έκθεση. Αυτά σημαίνουν ότι το τρέχον σύστημα λειτουργικά δεν, ε, επιχειρησιακά δεν είναι λειτουργικό και επομένως η ασφάλεια δεν είναι 100%. Ενώ όψη του τεράστιου προβλήματος δρομοκρατικών απειλών, όπως είπε και ο κύριος Πάτεν προηγουμένως, είναι σαφές ότι θα πρέπει αμέσως να πάυσουν θεωρήσεις που να ισχύουν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα αμέσως επαναλαμβάνω και να αντικατασταθούν από διμερείς θεωρήσεις από ε, έμπιστες χώρες. Τώρα να προσπαθείτε να ε, διορθώσετε κάποιες λεπτομέρειες του συστήματος δεν αποτελεί λύση. Χρειάζεται μια σε βάθος αναδιατύπωση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τελίτσκα ζήτησε να σας υποβάλει ερώτηση με μπλε κάρτα. Μια στιγμή να το ελέγξω. Okay, I think there's a seating issue. Who is wanting to raise the blue? Όχι, υπάρχει πρόβλημα της τις ε, έδρες. Ποιος ήθελε να θέσει την μπλε κάρτα, την επερώτηση με μπλε κάρτα. Κυρία Τζέμις, το δέχεστε. Ποιος όμως, κυρία Πρόεδρε, γιατί ε, δεν άκουσα καλά. Ο κύριο Στόιλερ. Όχι, δεν τη δέχομαι την επερώτηση με την μπλε κάρτα. Καλώς, ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη ομιλητριά μα για 1,5 λεπτό, η κυρία Γκραπίνη. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, φυσικά συμφωνώ και εγώ με την τροποποίηση του ελόγου κανονισμού που καθιερώνει ένα ενιαίο τύπο θεώρησης. Είναι απολύτως απαραίτητη η αναθεώρηση αυτή, όπως μας το δικαιολόγησε και η συγγήτρια με την οποία συμφωνούμε. Έτσι θα καταπολεμήσουμε τις παραποιήσεις, πλαστογραφίες, παραχαράξεις των αυτοκόλλητων ετικετών των θεωρήσεων. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο και ο ενιαίος τύπος θα μας το επιτρέψει. Πολλό δε μάλλον που οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυξάνονται και η κατάσταση της ασφάλειας ε, είναι δύσκολη. Θα πρέπει οι θεωρήσει να είναι ασφαλεί και να πληρούν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να γίνεται δύσκολη ή αδύνατη η πλαστογράφησή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι οι, σημαντι... οι σημερινές ε, αυτοκόλλητες ετικέτες θεωρήσεις δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια θεώρηση ενιαίου τύπου και για την ασφάλεια των πολίτων, αλλά και για την ισότιμη μεταχείρισή τους. Θεωρώ ότι οι συμπολίτε μου, αλλά και πολίτε άλλων χωρών που δεν ανήκουν ακόμη στο χώρο Σέγγεν, θα πρέπει να τύχουν ίδια μεταχείριση. Και μετά την υιοθέτηση τη τελευταία τροποποίηση του κανονισμού, πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο βήμα. Δηλαδή να καθιερώσουμε έναν ενίο χώρο έναν ενίο τύπο θεωρήσεων και ισότιμη μεταχείριση ενία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Σοροπέ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλούμε για ένα έγγραφο που αφορά τις αυτοκόλλητες ετικέτες των προξενικών θεωρήσεων και το θέμα δεν είναι αμφιλεγόμενο. Όλοι συμφωνούμε ότι οι ετικέτες αυτές οι αυτοκόλλητες θα πρέπει να είναι ασφαλείς και να μην επιδέχονται παραποίηση παραχάραξη. Γι' αυτό και συμφωνούμε με την πρόταση. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, οργανωμένο και μη. Υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα αφενός που ελπίζω να επαρκούν για να θωρακίσουν αυτές τις αυτοκόλλητες ετικέτες στις προξενικές θεωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κυκλώματα εγκληματικά που παραχαράσουν ε, επίσημα έγγραφα. Και μάλιστα αυτά τα κυκλώματα ασκούν ε, πολλές εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και εμπορία ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτές τις πτυχές και να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο στα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που διαχειρίζονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λεμπρετών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση. Το σύστημα Σέγγεν δυστυχώ ευνοεί αυτό το φαινόμενο γιατί αντικαθιστά τα εθνικά σύνορα με τα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση. που γνωρίζουμε ότι είναι τρίπια. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουν τουλάχιστον να περιορίσουμε το φαινόμενο. Οπότε αυτό κάνει αυτή η πρόταση, να αντικατασταθούν οι παλιές θεωρήσεις που εύκολα πάρει χαρά σε με μια άλλη πιο ασφαλή θεώρηση. Παρ' όλα αυτά, 22 χρόνια είχαμε έναν τύπο θεώρησης που βοηθούσε τις απάτες και πολλοί και εκμεταλλεύουν αυτή την κατάσταση για να μπουν παράνομα στην Ένωση. Τέλος πάντων, καλλιοργά αργά παρά ποτέ. Όμως πιστεύω ότι δεν θα αλλάζατε τίποτε εάν το εθνικό μέτωπο και η σύμμαχή του ε, δεν ε, ήταν εδώ στο Κοινοβούλιο τρία χρόνια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Συναδεινό. Η σημερινή αντίληψη περί ασφάλειας βασίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και απαρχιωμένες θεωρήσεις. Δεν αποδέχομαι εκπτώσεις στις υψηλότερες δυνατές τεχνικές προδιαγραφές προς αποτροπή της πλαστογράφησης και της παραποίηση εγγράφων θεώρησης απόλυτε βέβαια προποθέσει παραμένουν η καθολική συμφωνία συμμετοχή και έγκρισή του από τα κράτη μέλη του χώρου σέγγεν. αγνοείται όμω και μια κρίσιμη θεμελιώδη παράμετρο η κάλυψη αυτών των κενών δεν αποτελεί ικανή συνθήκη ή εγγύηση ώστε να περιοριστεί η δράση εκείνων των νομοκρατών, που ανατράφηκαν γενναιόδωρα αλλά δεν ενσωματώθηκαν και ριζοσπαστικοποιήθηκαν ανεξέλεκτα εντό τη ευρωπαϊκή επικράτεια. στο συγκεκριμένο τομέα οι προτινόμενε προσθήκε είναι απλώ ανεπαρκεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της σημερινής πραγματικότητας δεν είναι η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού είναι η κατάργηση της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην ένωση συχνά ως φτηνά εργατικά χέρια. αλλά τέτοιες πολιτικές μόνο εθνικιστικές κυβερνήσεις έχουν το σθένος και τη δύναμη να το πράξουν και θα το κάνουν να είστε σίγουροι. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Πίτσουλα για 1,5 λεπτό. Τα τελευταία χρόνια η πλαστογράφηση των αυτοκόλλητων ετικετών εμφανίστηκε σε αρκετά χώρα μέλη, σε αρκετές χώρες μέλη, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ασφαλές το ισχύον μοντέλο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο του 1995 που είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια της συνεργασίας στο χώρο Σέγγεν. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες προδιαγραφές. Η βελτίωση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων ε, είναι θεμελιώδη ζήτημα που αφορά και την προστασία των πολιτών. Και ε, είναι πρόσδεκτη η πρόταση αυτή γιατί πιστεύω ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας. Είμαι υπέρ της ανάπτυξης ε, θεωρήσεων ενιαίου τύπου με πιο ασφαλείς ετικέτες που θα εμποδίζουν ε, την παραχάραξή τους. Βέβαια, οι ασφάλειες ε, ε, οι απειλές στην ασφάλεια είναι σημαντικέ προκλήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και θα, θα προσδιορίσουν το χαρακτήρα της Ένωσης σε επόμενες δεκαετίες. οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι είναι όλο, και απα, όλο πιο απαραίτητη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αρχών ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και τις ε, χώρες ε, μέλη να συνεργαστούν καλύτερα, να ανταλλάσσουν καλύτερα τις απόψεις, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση της κατάστασης ε, των γειτονικών χωρών. Και επειδή η ασφάλεια είναι ο σημαντικός κρίκος της αλυσίδας, η σχετική συνεργασία στα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσόκα, για ένα λεπτό. Pazzesco pensare di raccontare ai cittadini europei, cittadini italiani στους Ευρωπαίους και στους Ιταλούς λέμε ότι με αυτόν τον ενίο τύπο θεώρησης δίθεν θα σταματήσουμε την τρομοκρατία και την ε, εισβολή των λαθρομεταναστών ε, ψηλά έτσι ο πήγης των ε, προσδοκιών έτσι λοιπόν φέρεστε σε Ευρωπαίους και σε Ιταλούς αν ήταν ηλίθιοι τα είναι δραματικά λέμε για 60.000 αποβιβάσεις λαθρομεταναστών γιατί αυτοί μετά οι 60.000 δεν ξέρουμε πού πήγαν γιατί εξαφανίστηκαν. 400% αυξήθηκαν οι Νιγηριανοί στη χώρα μας και έχει αποτύχει η πολιτική της κατάσταση στην Ευρώπη. Και έχουμε ένα εκατομμύριο που είπαμε θα επαναπατρίσουμε αλλά δεν έγινε τίποτα. Επομένως από εμάς περιμένουν να μπορούμε με τον ενίο τύπο θεώρησης γρήγορα να επισημαίνουμε τους λαθρομετανάστες, να τους επαναπατρίζουμε και αυτό θα έπρεπε να συζητούμε τώρα. Ο πρόεδρος και τώρα αρχίζει η διαδικασία Eye και ο πρώτος είναι ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο τύπος θεώρηση του Σέγγεν τώρα έχει, θεωρείται απαρχαιωμένος, οπότε θέλουμε ένα, ένα νέο τύπο για να υπάρχουν εγγύσεις μη παρχάραξης και πλαστογραφίας Επομένω, θα πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα γιατί έχουμε την απειλή τη τρομοκρατία. Εδώ έχουμε κενά όσον αφορά τον έλεγχο των θεωρήσεων. Επομένω, θα πρέπει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον έννοιο τύπο θεώρηση που έχει κάποια τεγκά χαρακτηριστικά το οποίο είναι πιο ασφαλή. Και ε, να υπάρχουν μέσα κατά τη παραχάραξη χωρί παρόλα αυτά να υπάρχει αυξημένο διοικητικό ε, κόστο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις πλαστογράφησης ε, πολλά κρατημέλη. Εδώ το λένε οι αρμόδιες ε, αρχές ε, και κυκλοφορούν πάρα πολλά πλαστά διαβατήρια. Επομένως θα πρέπει κατεπηγόντως κάτι να γίνει με αυτές τις απόρριτε τεχνικές ε, προδιαγραφές και σύντομα η σχετική νομοθεσία να εγκριθεί. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση επιχειρεί να αναθεωρήσει τον ε, ενιαίο τρόπο θεώρησης της βίζας προκειμένου όπως λέει να κλείσει τα παράθυρα για να μην υπάρχει δυνατότητα πλαστογραφίας. Όμως ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει τις πόρτες διότι έχει καταργήσει την βίζα για τους Κωσοβάρους. Δηλαδή στο Κόσοβο όπου είναι η σφυγγοφολιά πραγματικά των τζιχαντιστών η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταργήσει τη βίζα. Επομένως χωρίς βίζα αυτοί θα μπορούν να εισέρχονται. Και έτσι ο κίνδυνος τρομοκρατίας είναι αυξημένος. Και εμείς μιλάμε πώς εδώ θα κλείσουμε το παράθυρο για να μην γίνεται η πλαστογραφία. Όταν υπάρχει πλέον διγλωσία. Δεύτερον, έχετε καταργήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη βίζα για την Ουκρανία και μπορεί να εισέρχεται ο καθένας. Τρίτον, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την θεωρία των ανοιχτών θυρών. Ο κάθε ένας παράνομος μετανάστης έρχεται και μιλούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τροποποιώντας τη μορφή με την οποία γίνεται η ενιαία θεώρηση. μόνο όταν υπάρξουν εθνικά σύνορα μπορεί να καταργηθούν αυτές οι, οι ιστορίες που υπάρχουν με τους παράνομους που εισέρχονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα το λόγο στην κυρία την Επίτροπο. Σα ευχαριστώ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο του στο πολύ αυτό σημαντικό μέτρο της ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αυξανόμενο αριθμό των παραχαράξεων και παλαστογραφήσεων των αυτοκόλλητων ετικετών, Το θεωρήσω σε πολλά κρατημέλη. Ε, η αυτό, η αυτοκόλλητη αυτή ετικέτα που χρησιμοποιούνται, όπως μας λένε οι εμπειρογνώμονες, δεν είναι πια ασφαλής. Από την κυκλοφορία των πρώτων αυτών ετικετών προέκυψε η ανάγκη για αναθεώρησή τους να έχουμε νέα, ε, νέες αυτοκόλλητες ετικέτες πολύ πιο ασφαλής. Το κόστος της αγωγής των νέων αυτοκόλλητων ετικετών δεν θα υπερβαίνει το κόστος των παλιών ετικετών. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση της παραχάραξης εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη στιγμή που υιοθετηθεί το νέο μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της από όλε τις χώρες μέλη του Σέγγεν και από τις χώρες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να λάβουν μέρος και αυτές στην εφαρμογή του μέτρου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Κάουφμαν έχει το λόγο, η συγκήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εσά, κύριε Επίτροπε Επιθυμώ να ευχαριστήσω και όλες και όλους τους συναδέλφους που ε, συμμετέσχουν στη συζήτηση. Στο σύνολό της συζήτηση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που θεωρεί ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο τύπος των ε, προξενικών θεωρήσεων και όπως τονίσατε πολύ εξημών είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται εδώ στην κοινή μας Ευρώπη και ποιος παραμένει. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και βεβαίως πρέπει να ελέγξουμε από κοινού τα εξωτερικά μας σύνορα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Ευχαριστώ όλους και όλους τους συναδέλφους και πάλι για την καλή συνεργασία. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται πάλι το μικρόφωνο, απευθύνω έκκληση σε όλες τις χώρες μέλη μετά από το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου και μετά από τη σημερινή ψηφοφορία να σπεύσουν να εισαγάγουν το νέο ενίο τύπο θεώρησης και να μην εξαντλήσουν τους 15 μήνες της μεταβατικής περίοδου που κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικά μακρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κάουφμαν. Εδώ λοιπόν λίγη η συζήτηση και η ψηφοφορία.